θα ήλπιζα να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και ε, το επόμενο θέμα είναι αιτήσει ε, που μου έχουν γίνει για πολιτικές ομάδες, για μέτρα, για μέλη σε αντιπροσωπείες ε, για την ε, Νότιο Αφρική 2 ε, και ε, για την αντιπροσωπεία για το Παναφρικαϊκό Κοινοβούλιο Jim Higgins, Ευρωπαϊκή Ένωση Χιλή Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ, Ντι Φερνότικα Λόπε Φοντανιέ, ε, σχετικά με τις Ηνωμένε Πολιτείες Καρίμ Ζερίμπη και στην Ειδική Επιτροπή για, την το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά η κυρία Νικόλ Κι Νίλσεν. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση οπότε επιβεβαιώνονται και ε, διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 12. Ευχαριστώ.